αύξηση της ανάπτυξης επιτάχυνση αύξηση των θέσεων εργασίας υλοποίηση της στρατηγικής εε εξορθολογισμός και εξυγίανση της εταιρικής διακυβέρνησης διαφάνεια στην οικονομική διακυβέρνηση έλεγχος στα εθνικά στατιστικά δεδομένα μόνιμος μηχανισμός συνδιαχείρισης κρίσεων στην ευρωπαϊκή ένωση προς όφελο πάντα του ευρωπαίου πολίτη. η κρίση αφορά όλου και όχι μεμονωμένα τι χώρε που τη βιώνουν. αυτό που απαιτείται είναι κοινοτική αλληλεγγύη και συντονισμό δράσεων. ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μάντλενερ τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.